μεγάλη σημασία. Πρέπει να κατανοήσουμε όμω ότι χρειάζεται χρόνο για να επιτευχθούν και επομένω δεν θα πρέπει μονάχα να επικρίνουμε, θα πρέπει να βοηθούμε και την Ουκρανία να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή μα οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πίνκε Βιτσιούτε. Η κυρία Οβίερ έχει το λόγο.